Ευχαριστώ. Η κυρία Σαλτεμόζε. Ευχαριστώ πολύ. Onorevole Γκέτρουντ. Τζέσικα Γκέτρουντ. Πού είστε? Ωραία, δέχεστε, ευχαριστώ. Ράφαελ Γκλούξμαν. Πού είστε, ωραία. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Πάολο Μπόρκια. Ευχαριστώ πολύ. Κατερίνα Κονέτσνα. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Στεφάν Σεζουρνέ. Ονορεύολε Ιρένα Ιωβεβα. Ιρένα Ιωβεβα. Πολύ ωραία, ευχαριστώ και εσάς. Λοιπόν, ο κύριος David Ιβαν παίρνει το A και B. Η κυρία Σάλτε Μόζε το C, D Γκρουτ Γκρουτ-Ι έως G. Γκλούξμαν H έως K. Μπόρκια Λ Ελ-Μ. Η κυρία Κονέτσνα N έως R. Σεζουρνέ S έως T. Και Γιώβεβα U έως και Z. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ οι ψηφολέκτες ε, να έρθουν εδώ στο έδρανο της Προεδρίας, γιατί αν μπορείτε παρακαλώ να έρθετε. Και θα περάσουμε τώρα στη διανομή των ψηφοδελτίων και των φακέλων. Πριν ψηφίσετε, παρακαλώ να περιμένετε να κηρύξω την έναρξη της ψηφοφορίας και να ακούσετε τις συγκεκριμένε διευκρινήσεις. Οδηγίες χρήσης αν θέλετε. Για να ψηφίσετε παρακαλώ να σημειώσετε υπέρ με συν ή κατά με πλήν. Εάν ε, θέλετε να απόσχετε μπορείτε να αφήσετε ε, το ψηφοδέλτιο λευκό. Εάν θέλετε να διορθώσετε την ψήφο, να ζητήσετε νέο ψηφοδέλτιο θα σας τη δώσει κλητήρα σε αντάλλαγμα του λανθασμένου ψηφοδελτίου, το οποίο θα καταστραφεί. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε επιγραφή ή οποιαδήποτε ένδειξη στο ψηφοδέλτιο, εννοείται ότι θεωρείται άκυρο. Θα πρέπει να το διπλώσετε στα τέσσερα και να το βάλετε στο φάκελο. Έχετε στη διάθεσή σας ε, και ε, καμπίνες, ε, αν κάποιος επιθυμεί να ε, τις χρησιμοποιήσει. Μπορείτε να πάτε ε, στην αντίστοιχη κάλπη που αντιστοιχεί στο επιθετό σας. Θα πρέπει να δείξετε ή κάποιο έγγραφο ταυτότητας ή το μπάντ σας στο ψηφολέκτη πριν ψηφίσετε. Allora, scusate a tutte. Λοιπόν, έχουμε ψηφολέκτη σε όλες τις κάλπες. Alors, ε, οι ψηφολέκτες θα ψηφίσουν μετά το πέρας της ψηφοφορίας. Άρχεται η ψηφοφορία. Ο κύριος Μπόρκια θα πρέπει να πάει στην κάλπη L έως και M. Παρακαλώ. Ευχαριστώ.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, ψηφίζετε όλοι. Ψήφισαν οι ψηφολέκτες. Νομίζω ναι. Επομένως, πέρα της συνεδρίασης, οι ψηφολέκτες θα πρέπει να πάνε στην αίθουσα R11 για να ε, γίνει η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και το άνοιγμά τους και ως συνήθως το κουδούνι θα ανακοινώσει την ε, συνέχεια της συνεδρίασης. Διακόπτεται η συνεδρίαση, θα το δείτε και στις οθόνες.